Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε ξεκινούμε με την ψηφοφορία για την διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη. Καλώς ορίζω τους συναδέλφους της Ιδρύα και τον Πρόεδρο. Έχετε τις κάρτες σας όλοι, ελπίζω. δεν μπορείτε να ψηφίσετε χωρίς κάρτα. Διανατάσσεως της χειρός δεν είναι δυνατή η ψηφοφορία. Και Κραμά. Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας μου, σας ενημερώνω ότι διαμαρτυρόμεθα συμμετέχουμε με επιφύλαξη, διότι οι κανόνες αλλάζουν συνεχώς. Χθε μας έδωσαν κατάλογο ψηφοφορία με τροπολογίες που δεν συζητήσαμε. Συζητήθηκαν οι συμβαστικέ ψηφοφορίε μεταξύ των δύο μεγάλων ομάδων, μόνο. Η τροπολογία, μία τροπολογία που κατέθεσαν τέσσερι άλλε ομάδε δεν συζητήθηκε. Αλλάζουν διαρκώ οι κανόνε ανεξέλεγκτα. Χθε του συντονιστέ. Προτείναμε χωριστή ψηφοφορία. Τρεις συντονιστές υπερψήφισαν, τέσσερις κατά, είχαμε μία αποχή. Και μας είπαν χθες ότι, ξέρετε, έστω και με τρεις υπέρ, απορρίπτεται η συμβαστική. Μετά είπαμε όχι στις ε, χωριστές ψηφοφορίες και μετά η Ήτρε ε, ζήτησε ξανά χωριστή ψηφοφορία στο παράδειγμα, Το απόγευμα άλλαξαν πάλι όλα αυτά, όχι στη χωριστή ψηφοφορία. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε έτσι. Η άποψή μας δεν έγινε ακουστή, το θεωρώ απαράδεκτο. Χθε πήραμε τον κατάλογο ψηφοφορία σε μία μονογλώσσα βασική παραβίαση των κανόνων εργασία. Διαμαρτυρόμεθα λοιπόν, δεν συμφωνούμε, ε, συνεχίζουμε να συμμετέχουμε, αλλά θα προβούμε σε κάθε ε, είδου παρήθευση για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι νόμιμα. Κύριε Κράμερ, λέει ο πρόεδρο. ε, κατανοητό σημειώνω, θα επανέλθετε αργότερα και ξεκινούμε με την ψηφορία. Διακόπτη. Πρόεδρε. Έχουμε 69 συμβαστικέ πληροφορίε από των οποίων πρέπει να ψηφίσουμε 85 σελίδε. Δεν ξέρω εάν οι κανόνε της πολυγλωσσίας τηρούνται, εν προκειμένου. Πρόεδρος, μου είπαν ναι, μου λένε ναι. Η γραμματεία μου λέει ναι, η γραμματεία της ΙΤΡΕ. Πολύ ωραία. Οπότε προχωρούμε με βάση αυτά και ξεκινούμε με την ψηφοφορία για τον μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη. Βάλιεν και άλλοι Να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, να δω αν έχουμε απαρτία, ηλεκτρονικός έλεγχος και οι δύο επιτροπές βεβαίως πρέπει να έχουν απαρτία, οπότε ελέγχουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. ψήσαν όλοι. Ο καθένας θα πάει στη θέση του παρακαλώ για να ξέρουμε ποιος κάθεται πού, από ποια επιτροπή. Ε, φαίνεται ότι εδώ μια τρίτα δεν ε, δουλεύει. Πέρας ψηφορία η τεχνική να το φροντίσουν παρακαλώ. Είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, ξεκινούμε άρθρο 1. Κάνω τα χέρια σας, δεν χρειάζεται. Okay, rapporteur ready, Ines. Έτοιμοι οι συγητές. Ines. Λοιπόν, πώς θα προχωρήσουμε. Ξεκινούμε έναν μαραθώνιο κυρίε και κύριοι. Άρθρο 1, συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο κύριος Τόμασον υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 2.30. Επόμενη. Συμβαστική 1α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.35 προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2, 28 ε, με συγχωρείτε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σημειβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Στη σελίδα 5. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 263. 263 προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 272 προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2,78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπή Προπολισμών 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 και οι 2,80 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,84 προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.97 η κυρία Τίκαου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 305. Με συγχωρείτε λέει ο ε, έχω την 9. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα είναι 305 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 306 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 307 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3-10 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρία εικοσιδίο. Τρία προσθήκη για το διοξείδιο του άνθρακα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, έναρξη ψηφοφορίας, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 322. Για την 322 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι, πέρας. εγκρίνεται με σαφή πλειοψηφία. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία στο τέλος της προηγουμένης υπάρχει καμία αντίρρηση για την κατάθεση προφορικής τροπολογίας υπάρχει άρα δεν γίνεται δεκτή. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 οι επόμενες δύο καταπιπτούν λόγω της 43. Συμβαστική λοιπόν 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. πέντε. Θα τη βρείτε. Περιμένω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 349 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.55 προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχή. Απορρίπτεται. Πάμε πιο κάτω. Στην 370. Στη σελίδα 18 στο δικό μου έγγραφο τουλάχιστον. 370 προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 συμβαστική 20 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφορίας για την συμβαστική 20. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. 353 με την προσθήκη των ε, λέξεων ενεργειακή απόδοση. Ο κ. Τέμις, 353 υπέρ. Κατά. Απόδοση. Απορρίπτεται. Ε, λόγω της συμβαστικής ε, το υπόλοιπο κείμενο καταπίπτει. Η συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.88 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστ. 57. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 390 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ε, παρακαλώ. Να το ξαναδούμε. Ήρθε 390 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σεφώς. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 395 προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 399. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 396 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 397 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 398 και οι 400 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 401 προφορική, υπάρχει αντίρρηση για την υποβολή, υπάρχει μια αντίρρηση, άρα θα τη συζητήσουμε. 401 χωρίς την προφορική, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι, 23ο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 402 και 3 ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος 402 και 403, έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Το έλκ κέρδισε ένα σωρό. Α, μισό λεπτό. Μπορείτε να κλείσετε το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Ε, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, λοιπόν. Ρέτζι 21 και προπολογισμό 20 ταυτόσιμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 των εισηγητών υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 405 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 των εισηγητών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Εγκρίνεται. 404 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 406 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 407 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 408 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 409 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός 24 Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε και την συμβαστική 25, λίγες σελίδες πιο κάτω. Συμβαστική 25 είναι στη σελίδα 27 στο δικό μου το κείμενο, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω σε τι σελίδε είναι του ΕΛ των φιλελευθέρων. πάντων 25 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Τώρα έχουμε και τη συμβαστική 26 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 27, να το βρω ένα λεπτό, νάτινα, νάτινα, λέει ο Πρόεδρος, υπέρ, της 27, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 28, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 476, υπέρ, καταπεπτή, ρωτάει ο Πρόεδρος. Πού είμαστε, λέει ο πρόεδρο. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, 71, 71. Είμαστε στην τροπολογία 71. Η 476 καταπίπτει λόγω συμβιβασμού. 71, πού είναι το 71, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην ε, συμβαστική 29. Όχι, ο κύριος Γκρότ διαδικαστικό. Η 483 είναι ταυτόσιμη με την 71 και δεν το είπατε, Πρόεδρε. 483 ταυτόσιμη με την 71 και δεν το είπατε. Ναι, λέει Πρόεδρος, σωστά. Είναι ταυτόσιμες. Είναι ταυτόσιμες. Είναι αλήθεια αυτό. Τέλος πάντων, συμβαστική 29. Ε, πάντως εγκρίθηκε έτσι δεν είναι. Ωραία. Συμβαστική 29. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Κατά, εγκρίνεται. Πέντε δεκατέσσερα προσθήκη. Υπέρ. 5-14. Ε, Μάκ, νομίζω είσαι υπέρ της ε, τροπολογίας σου, έτσι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 498. Ξέρετε που είμαστε όλοι. Έχετε βρει το δρόμο σας. Ωραία. 498. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 23. Το τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ρέτζι 23. Πέμπτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ρέτζι 24. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 520 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 521 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 524 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 524 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. Τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε την 523 και την 572 μαζί. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Θα το λέξουμε και αυτό ηλεκτρονικά. 523 και 572 άρχεται η ψηφορία. Όχι. Όχι. Ψηφίσατε πέρα της 523. Καταπίπτει, αν θετική 24, όχι, αλλά τώρα καταπίπτει με το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία. Τροπολογία 79 υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. 525 κυρία Βίλ υπέρ. Κατά αποχέ, απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. της προπολογισμών 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 527 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 526 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα ελέξουμε αρχίζει η ψηφοφορία για την 526 Ψηφίσατε όλοι. Το ΕΛΚ έχει υπερβολικά μεγάλο αριθμό. Ό, όχι, εντάξει, εντάξει, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία, πέρα τη πληροφορία και εγκρίνεται. «81». Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 529 και 530 καταπίπτουν. «531» λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 32, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27, Ρέτζι, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 συμβαστική 33 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 και 49 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 550 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 547 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ...551 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, ...552 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 553 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 555 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 562 προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 563 και 564 είναι ταυτόσιμες ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 566 565 5 ταυτόσιμη με την 563 και 564 οπότε 566 της κυρία Wills υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά άποχες άλλη μια φορά παρακαλώ 95 υπέρ έτσι μπράβο κατά άποχες εγκρίνεται 567 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η Reggie 28 καταπίπτει. Οπότε πάμε στην 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε τώρα τη συμβαστική 36 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 571 υπέρ. Κατά. Άποχες να ελέξουμε για την 571 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Μάτιο και Γιώργο, ναι, να έχετε τις κάρτες σας. Εντάξει, όλα εντάξει, πολύ ωραία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Ρέτζι 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Την Ρέτζι 30 αρχίζει η ψηφοφορία. Γιώργος, παρακαλώ, μπορείς να κοιτάξεις τι γίνεται. Ναι, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 573 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 574 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 574 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 ε, από πρόεδρος ήταν 5. 576 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 32 καταπίπτει. 577 και 578 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 37. Υπέρ. Ξαναρχίζουμε, λέει ο πρόεδρος. Συμβαστική 37. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 582. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 της Ρέτζη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Συμβαστική 38. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Προπολογισμών 30. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 584 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 585 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 586 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 και 587 είναι ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39α υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 39β ένα λεπτάκι 39β ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, αλφαβητικά πάμε λέει ο πρόεδρος αλφαβήτα γάμα δέλτα ε 39 ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 ζήτα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 ήτα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39Θ θήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 γιώτα υπέρ. όχι, όχι, λάθος, λάθος, λάθος. Ε, ναι, ναι, ναι, τρέχω πολύ ο πρόεδρος. 39 γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...39 καί στα αγγλικά. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Αλλά θα ελέξουμε. Θα ελέξουμε για την 39 K στο αγγλικό. Ωραία. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. εγκρίνεται. One fence at a time, Georges. One fence at a time. Ένα-ένα. Ένα-ένα με τη σειρά, Γιώργο. Now we got a compromise. Συνεχίζουμε. Συμβαστική 40. Το βρήκατε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Περνάμε στην 734 προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 742 προς την Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Συμβαστική. Α, Ρέτζι. Ρέτζι 1. Λέω πρόεδρος. Υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Budget 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 είναι γλωσσικού χαρακτήρα, χαρακτήρα. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 44 γάμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 και 137 ταυτόσημε υπέρ. Κατά. εποχέ, Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. εποχέ. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 δέλτα. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. 44 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτσι 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 151. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Και πάλι. Υπέρ της 150. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εντάξει, να ελέγξουμε την 150. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίτεται. Συμβαστική 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 είναι προσθήκη. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Όχι, εντάξει, θα το ελέγξουμε. 154 ως προσθήκη. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Εντάξει. Λύθηκε το πρόβλημα. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Εντάξει, με μικρή διαφορά. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 157. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 46. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 160. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 160. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Α, να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 174, έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 49, επέ. Κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 να είναι σαφές 178 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Βάτζετ, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ελεκτρονικό έλεγχο τη 182. Νομίζω ότι έχει περάσει, αλλά να το δούμε. Έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 50α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 194. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 194. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2-10-2-11 ταυτόσιμες. να Θέλετε να ελέγξουμε την 209. Εντάξει, έναρξη. περα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2-10 και Ρέτζι 11 ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. αποχε Εγκρίνεται. 2.12 υπέρ. Όχι. 2-11 πρώτα. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τώρα Τώρα 2-12 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 52 συμβαστική 52 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 2.17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.18 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ρέτζι 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.21 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος της 2.21 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Έγκρινεται λοιπόν. 22 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχο. Γιατί πολύ λίγοι ψήφισαν. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, ε, Εγκρίνεται. 2.27 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 2.28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Budget 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Budget 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Να υπενθυμίσω ότι με τους νέους κανόνες έκθεσης Κορόρες ε, θα υπάρχουν τρεις ψηφοφορίες γι' αυτό. Ψηφίζουμε επί της ε, πρότασης όπως έχει τροποποιηθεί, μετά την νομοθετικό ψήφισμα και μετά τις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις. Εντάξει, ωραία. Νομοθετική πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί με ηλεκτρονικό έλεγχο. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 80 υπέρ, 8 κατά, 5 αποχές. Υιοθετείτε το νομοθετικό ψήφισμα έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Πέρας. 81 υπέρ, 8 κατά, 5 αποχές. Εγκρίνεται και πάλι και ψηφίζουμε τώρα για την διοργανική διαπραγμάτευση, η έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 86 υπέρ, 6 κατά, 2 αποχές. Να συγχαρώ τους τρεις εισηγητές λοιπόν. And Να δώσω το λόγο τώρα στην, στο, στην πρόεδρο Σαρτόρη. Μην φύγετε ακόμα, κυρίε και κύριοι. Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τους συγγητέ για αυτή τη θαυμάσια δουλειά που απέδειξε ότι μπορούμε να εργαστούμε καλά και να συνεργαστούμε σωστά με μια διαδικασία έτσι φορτωμένη και δύσκολη όπως η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Θα συνεχιστεί η δουλειά μας με τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και ελπίζω και αυτή η διαδικασία θα είναι εξίσου επικοδομητική. Καλό τους συναδέλφους τη Σύντρε να πάνε στη 5 B001 ε, που θα συνεχίσουμε τις δικές μας εργασίες. Ευχαριστώ και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε διάλειμμα 10 λεπτά τώρα. και θα προχωρήσουμε με την επόμενη ψηφοφορία μας. Ευχαριστώ.